Good Καλή σας μέρα. Δεν είμαστε και πολύ σήμερα, αλλά ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε. Παρόλο που πολλοί συνάδελφοι ίσως κόλλησαν σε μποτιλιάρισμα, στο δρόμο τους προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάποιοι δεν θα Προφθάσουν να έρθουν εγκαίρως, αλλά αυτό δεν, θα πρέπει να μας εμποδίσει να ξεκινήσουμε στην πρώτη μας συζήτηση που θα κρατήσει μισή ώρα και αφορά τη συμφωνία, του το σημείο 7, Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβατικής Συνομοσπονδίας για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων για την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως ό,τι αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος και για την διαπίστευση παρόχων ε, εγκληματολογικών υπηρεσιών που πραγματοποιούν εργασίες εργαστηρίου. Η συγκίτρια της έκθεση είναι η κυρία Μετσόλα, που επίσης δεν πρόλαβε να έρθει. Είναι καθοδόν. Αλλά για την παρουσίαση του σημείου 7 θα την αντικαταστήσει η συνάδελφός της η κυρία Dupont. Και φυσικά θα έχουμε ένα γύρο συζήτηση με τους κοιόδης συγγητές. Μάλιστα, για το σημείο 7 προβλέπεται κοινή συζήτηση με το σημείο 8 που αφορά ένα παρεφερές θέμα το οποίο επίσης έχει αναλάβει η κυρία Μετσόλα. Το σημείο 8 αφορά τη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν. Το αντικείμενο όμως είναι το ίδιο, οπότε και οι σκιώδεις είναι οι ίδιοι. Γι' αυτό και προτείνω να γίνει κοινή συζήτηση των σημείων 7 και 8. Θα ακούσουμε την ενημέρωση από τον κύριο Ντυπών και μετά θα μας πούν τη γνώμη τους οι σκιώδεις ηγητές. Πριν σας ανακοινώσω την προθεσμία ή τις προθεσμίες των διεκθέσεων για την υποβολή τροπολογιών. Κύριε Ντυπών, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φυσικά δεν είμαι η Ρομπέρτα Μετσόλα. Θα προσπαθήσω όμως να την αντικαταστήσω επάξια. Οι δύο ε, εκθέσει τη είναι απλέ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να διερευνήσει τη δυνατότητα να δώσει τη συγκατάθεσή του για δύο ξεχωριστέ συμφωνίε μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελβετία αφενό και Ευρωπαϊκή Ένωση και Λιχτενστάιν αφετέρου για την εφαρμογή κάποιων διατάξεων τη απόφαση του Συμβουλίου για την καταπολέμηση ε, τρομοκρατία και διασυνοριακού εγκλήματο και ε, τη απόφαση πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη διαπίστευση των παρόχων εγκληματολογικών υπηρεσιών που παρέχουν εργασίε εργαστηρίου. Φυσικά μα ενδιαφέρει η αναβάθμιση τη ασφάλεια Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα τρόπο που το κάνουμε είναι να διευκολύνουμε ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα επιβολή νόμου με τι αρμόδιε αρχέ. Γιατί δεν μπορεί μια χώρα μόνη τη να σταματήσει το διασυνοριακό έγκλημα που δεν γνωρίζει σύνορα. Ε, γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε ενίσχυση των, ε, της συνεργασίας των ε, υπηρεσιών επιβολή του νόμου ε, για την καταπολέμηση τρομοκρατία και διασυνοριακού εγκλήματο. Γι' αυτό και έχουμε τι δύο συμφωνίε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελβετία και ε, Στάιν για την ε, ανταλλαγή δεδομένων σχέση με την ανάλυση κάποιων στοιχείων, στοιχείων ταυτοποίηση και καταγραφή. Και γίνεται πληρούνται οι προποθέσει από τι δύο χώρε για την ανταλλαγή τέτοιων στοιχείων. Οπότε η σύσταση τη της τη κυρία Μετσόλα είναι να δώσουμε τη συγκατάθεσή μα στη συνένεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη σύναψη των δύο συμφωνιών. Ευχαριστώ. Θα ακούσουμε τώρα τους σκιώδη ηγητέ. Ο κύριο Μορένο Σάντζε είναι ο σκιώδη ηγητή των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλημέρα σα. Η ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποστηρίζει αμέριστα τις ε, δύο εκθέσεις, γιατί θεωρούμε ότι είναι σημαντική η αστυνομική συνεργασία. Δεν θα, μπορούν, δεν θα πρέπει τρομοκράτες και οι εγκληματίες να κυκλοφορούν ανενόχλητα από τη μία χώρα στην άλλη. Γιατί είχαμε προβλήματα με την τρομοκρατία της Αλκάιδα, των τζιχαντιστών. Είναι σημαντικό να αποτρέψουμε ε, να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία και το διασυνοριακό έγκλημα και οποιαδήποτε αναβάθμιση συνεργασία ε, είναι ευπρόσδεκτη. Γι' αυτό και συμφωνούμε με την συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Εγώ αντικαθιστώ σήμερα τον συνάδελφο Άντωνη Χουκ, που επισκολύεται. κολλιέται. Πάντως, και ο Άντωνη συμφωνεί με την παροχή συνένεση <clears throat> εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στι δύο συμφωνίε. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα του Σκιώδου Σιγητού. Η καταπολέμηση τρομοκρατία και διασυνοριακού εγκλήματο είναι ύψιστη προτεραιότητα και των Ευρωπαίων πολιτών, όπω δείχνουν οι δημοσκοπήσει. Γι' αυτό χαιρετίζουμε τη συμφωνία των αποφάσεων ε, αυτών και θα πρέπει να εξασφαλιστεί καλύτερη διαλεύκανση των ε, εγκλημάτων με ενίσχυση τη αστυνομική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των δύο χωρών. Επίσης, έχουμε την ε, αναβάθμιση της ε, συνεργασίας ό,τι αφορά τη διαπίστευση παράχωρων κλιματολογικών υπηρεσιών, κάτι που θα διευκολύνει τη διαλεύκαση εγκλημάτων. Σίγουρα είναι διασυνοριακό ο χαρακτήρα του Διεθνού Οργανωμένου Εγκλήματο και δεν γνωρίζει σύνορα ούτε κατά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό χαιρετίζουμε τη δυνατότητα που προσφέρεται στα κράτη-μέλη να έχουν πρόσβαση στι εθνικέ βάσει δεδομένων τη Ελβετία και του Λιχτενστάιν, σε ό,τι αφορά το DNA, δακτυλοσκοπικά στοιχεία και στοιχεία ε, ταυτοποίησης. Ε, πάνω από 4.000 ε, συμμορίες ε, ενεργοποιούνται διεθνώς και βρίσκονται υπό έρευνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να καταπολεμηθούν αυτά τα φαινόμενα, είναι σωτική σημασία η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου. Και μάλιστα ε, το Μάιο ολοκληρώθηκαν οι συμφωνίε ε, με το Λίχτενστάιν και την Ελβετία και ευχαριστώ την κυρία Μετσόλα, την εισηγήτρια, για τη δέουσα προσοχή που αφιέρωσε στι δύο αυτέ σημαντικέ συμφωνίε. Ευχαριστώ και τώρα για του πράσινου. Μάλλον όχι, δεν βλέπω. Βλέπω τον κύριο Κόφουντ ε, για την ομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εμένα δεδομένη σε έλλειψη απαρτίας που έχουμε, θεωρώ πολύ παράδοξο το ότι συνεδριάζουμε παρόλα αυτά με τόσους λίγους, λίγους συναδέλφους. 6, 8, 10 είμαστε το πολύ. Πού είναι οι υπόλοιποι, γιατί δεν ήρθαν. Δεν ξέρω, έχουν άλλες παράλληλες συνεδριάσεις. Νομίζω ότι είναι πραγματικά παράλογο, αλόκοτο θα έλεγα, να συνεδριάζουμε τρεις και ο κούκος. Και απαράδεκτο κατά τη γνώμη μου, να συνεδριάζουμε ενώ δεν έχουμε απαρτία. Δεν έχω τίποτα να πω για τις δύο εκθέσεις. Ευχαριστώ. Δεν είσαι σκιώδης ηγητής, έτσι. Δηλαδή συχνά ε, έτσι μαθαίνουμε να δουλεύουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το έχω δει χιλίε φορέ. Ε, παραπονιούνται κάποιοι για την απουσία. Ε, δεν φταίει κανεί. Και μην κατηγορείτε του παρόντε. Γιατί αυτοί είναι εδώ τουλάχιστον. Πρέπει λοιπόν να εξηγήσουμε ε, στην κοινή γνώμη ότι καμιά φορά οι βουλευτές είναι αλλού. Δεν φταίει κανείς. Αλλά τέλος πάντων. Ε, είμαστε εμείς εδώ για να συνεχίσει η δουλειά μας. Σκιάστε λοιπόν. Αυτά για το πρώτο σημείο της ημερησίας διάταξης. Αρκετά. Το είχαμε προγραμματίσει μέχρι τις 9.30. Αν υπάρχει κάποιο σχόλιο από την βασική συγκίτρια του ΕΛΚ. Έχετε να προσθέσετε κάτι, όχι. Καμιά φορά η Κομισιόν θέλει να πει κάτι, όχι. Μάλιστα. Οπότε να υπενθυμίσω στους βουλευτές ότι επιτρέπεται να μιλήσουν μόνο σύμφωνα με το άρθρο 105 και 104 οι συγητές και οι συγητές. Οπότε η προθεσμία είναι στις 14 Νοεμβρίου, 6 ώρα το απόγευμα και η ψηφοφορία θα γίνει 2 Δεκεμβρίου. So, we've got a second Έχουμε και ένα άλλο θέμα που έχουμε προγραμματίσει σε 9.30 ώρα. Europol έχουμε μια παρουσίαση των Διευθυντή Επιχειρήσεων ε, της Europol 9.30 ε, ώρα. 9.30 ώρα δεν έχει πάει. Διάλειμμα ο λίγων λεπτών. Και μετά τα ξαναλέμε. Εντάξει, για καφεδάκι. Ευχαριστώ. Και σας ευχαριστώ για την κατανόηση. Ε, εντάξει, δεν είναι ευχάριστο να μην έχουν έρθει οι συνάδελφοι. Τι να κάνουμε. Ο Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε. Περνάμε στο δεύτερο σημείο της της διάταξης που αφορά την αξιολόγηση των απειλών όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα στο διαδίκτυο που πραγματοποιεί η Ευρωπόλ για το 2019. Θα μας κάνει την παρουσίαση ο κύριος Βιλ Βαν Χέμερτ, που είναι αναπληρωτή διευθυντή επιχειρήσεων της Ευρωπόλ. Καλώ ήρθατε κύριε Φανχέμερτ. Στις 9 Οκτωβρίου φέτος η Ευρωπόλ υιοθέτησε την έκθεση αξιολόγηση απειλών για το 2019, την IOCTA, όπως λέγεται. Η έκθεση αυτή αξιολογεί το τοπίο απειλών για το οργανωμένο έγκλημα στο διαδίκτυο και επικεντρώνεται σε βασικές απειλές τεχνητή νοημοσύνη, νέες ε, τεχνολογίες είναι πανταχού παρούσες. Οι αστυνομικές δυνάμεις βέβαια αντιμετωπίζουν προηγούμενες αλλά και νέες απειλές που προέρχονται κυρίως από γνωστά τροτά σημεία σε, στις υπάρχουσες τεχνολογίες. Καλώς ήρθατε κύριε Φανχέμερτ και εσείς και το επιτελείο σας και περιμένουμε να μας εξηγήσετε την έκθεση της ε, Ευρωπόλ για να μπορέσουμε στη συνέχεια να τη συζητήσουμε. Το σημείο αυτό θα συζητηθεί την επόμενη ώρα, μέχρι τις 10.30, δηλαδή μετά την παρουσίαση του κυρίου Φανχέμερτ. Θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Είναι τιμή για εμένα να παρευρίσκομαι για άλλη μια φορά στην Επιτροπή Θεμελιωδών Ελευθεριών για να σας παρουσιάσουμε σε συνεργασία με τους συναδέλφους μου την έκθεση ΑΕΟΚΤΑ. Είμαστε όλοι λοιπόν πολύ ευτυχεί που θα μπορέσουμε να σα κάνουμε αυτή την παρουσίαση και να απαντήσουμε στι ερωτήσει σα. Τις επόμενες, επόμενα 15-20 λεπτά θα σα παρουσιάσω την έκθεση ΑΙΟΚΤΑ και κάποιε από τι συστάσει τη. Βλέπετε και στην οθόνη σας η ΑΕΟΚΤΑ είναι μία από τις εμβληματικές εκθέσεις που προετοιμάζει ε, ετησίως η Europol. Είναι μια στρατηγική έκθεση για την κατάσταση στο ίντερνετ και το κύβερνο έγκλημα. Είναι μια αξιολόγηση η οποία βασίζεται στις ε, επιχειρήσεις ε, των ε, διοκτικών αρχών, αλλά επίσης λαμβάνουμε υπόψη μας και πληροφορίες από τα άλλα υπουργεία που ασχολούνται με το θέμα και πανεπιστημιακούς. Προσπαθούμε να εντοπίσουμε τις τρέχουσες επιλές, αλλά επίσης και τις τάσεις που διαπιστώνουμε στις ε, διάφορες έρευνές μας και να καταλήξουμε σε συστάσεις, σε προτάσεις προς εκείνους που λαμβάνουν τις αποφάσεις, δηλαδή εσάς. Σε όλα τα επίπεδα, είτε πρόκειται για το στρατηγικό επίπεδο, το επίπεδο πολιτικής ή και το επιχειρησιακό. Δεν αξιολογούμε μόνο λοιπόν τις απειλές, αλλά Επίσης προσπαθούμε να αναδείξουμε και κάποιες ευκαιρίες και κάποιες ε, επιτυχίες που σημείωσαν οι διοκτικές αρχές. Και στο τέλος της έκθεσης προσπαθούμε να προβλέψουμε και λίγο τι θα μας ε, επιφυλάσσει το μέλλον. σε σχέση λοιπόν με την αξιολόγηση απειλών, εάν έπρεπε να περιγράψω με μία λέξη το κυβερνοέγκλημα θα έλεγα τη θρασίτητα. Δηλαδή ότι όλο και περισσότερο ε, βλέπουν ε, τις διαφορές ευκαιρίες, αλλά και όλα τα άλλα που βλέπετε. Dark Web, 5G, ε, GDPR, όλα αυτά είναι μέρος της αξιολόγησής μας επόμενη διαφάνεια. Λοιπόν, αυτό το οποίο έχει αλλάξει και είναι συμβολικό εάν συγκρίνεται την πρώτη σελίδα της προηγούμενης έκθεσης με την καινούρια έκθεση. Στα αριστερά το 18 βλέπετε ότι εστιάζαμε στον εγκληματία, τον δράστη. Τώρα είναι περισσότερο ένα θέμα νοοτροπίας για το πώς ε, οι κυβερνοεγκληματίες εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες που τους δίνει η τεχνολογία. Τα σημαντικότερα συμπεράσματα είναι ότι οι επιθέσει με μεκά είναι πιο στοχευμένες, πιο επικερδεί και τελικά και πιο βλαπτικές για την κοινωνία μας. Κάτι το οποίο επίσης αυξάνεται είναι το πώ καταφέρνουν να πλήττουν τα email επιχειρήσεων και καταφέρνουν έτσι να αποσπούν χρήματα μια νέα μορφή λοιπόν, ισχυρότερη μορφή κυβερνοεγκλήματος. Το κομμάτι επίσης που αφορά παιδεραστία αυξάνεται συνεχώς και αποτελεί μεγαλύτερη πρόκληση για τις διοκτικές αρχές και γίνεται πιο δύσκολο επειδή και οι νεαροί παράγουν από μόνοι τους τέτοιο υλικό. Κάτι άλλο θετικό νομίζω είναι ότι έχουν κατέβει αρκετές ε, τέτοιες αγορές ε, στο μαύρο διαδίκτυο όπως η Wall Street Market και άλλες, ε, κάτι το οποίο το έχουν αποσταθεροποιήσει αρκετά. Κάποιοι πολιτές δηλαδή έχουν εξαφανιστεί εντελώς ή έχουν φτιάξει μεμονωμένα μαγαζιά και εξαφανίζονται διάφορες αγορές και χρησιμοποιείται επίσης και η κρυπτογράφηση ως βασική υπηρεσία. Βλέπουμε επιθέσεις denial of service ε, με ένα στοιχείο εκβιασμού. Επόμενη διαφάνεια. Στις ε, οριζόντιες τώρα τάσεις ε, βλέπουμε αυξημένη χρήση της κρυπτογράφησης. Επίσης έχουμε και τα κρυπτονομίσματα και την ανωνυμία στο διαδίκτυο, κάτι το οποίο καθιστά πάρα πολύ δύσκολο για τις ιδιοκτικές αρχές να έχουν πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα. Και καμιά φορά είναι σχεδόν αδύνατο. Και η δεύτερη οριζόντια τάση είναι ότι πλέον τα πάντα αφορούν τα δεδομένα. Τα δεδομένα ως ε, ένα υλικό εμπορεύσιμο ως στόχος ή ως ε, εργαλείο ή ένας τρόπος να γίνει αναγνώριση. Για εμάς έχουμε τρεις προκλήσεις. Ε, πρώτα απ' όλα η πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα στο πλαίσιο ερευνών, η διαχείριση των μαζικών δεδομένων και τέλος να τα χρησιμοποιήσουμε στις έρευνες. Ε, θα επανέλθω σε αυτά λίγο αργότερα. Επόμενη διαφάνεια. Αυτές είναι οι κατηγορίες ε, που αναφέρουμε στην έκθεση. Αν μπορώ να σας δώσω κάποιες λέξεις. Στο κυβερνοέγκλημα βλέπουμε τα λιτρισμικά, επιθέσεις όπως είπα, την άλλο service, επιθέσεις ε, στην ε, υποδομή και βεβαίως υπάρχει και ο βανδαλισμός των site για τις απάτες ε, πληρωμών. Εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με τις πιστοτικές ε, κάρτες, αλλά και στα ATM. Με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή να υποκλέπτονται τα στοιχεία των καρτών. Επίσης βλέπουμε να γίνεται η πρώτη χρήση τεχνητής νοημοσύνης από τους ε, εγκληματίες, δηλαδή προσπαθούν να μιμηθούν ε, την φωνή διευθυνών των συμβουλών. Επίσης ε, έχουμε κοινωνική, μηχανική, δηλαδή εξακολουθεί ο άνθρωπος να είναι ο ασθενέστερος κρίκος. Για το έγκλημα ως υπηρεσία έχουμε τα βαποράκια χρημάτων, αυτοί οι οποίοι έχουν τους λογαριασμούς στους οποίους πάνε τα λεφτά, κρυπτονομίσματα επίσης ε, αποτελούν πλέον στόχο των εγκληματιών. Βλέπετε εκεί ότι ε, πηγαίνουμε προς μια ψηφιοποίηση. Για ζητήματα παιδεραστίας ε, στο διαδίκτυο έχουμε την διανομή του υλικού αλλά και την άγρα των παιδιών ε, στο διαδίκτυο και όπως σας είπα υπάρχει και το υλικό το οποίο παράγουν οι ίδιοι οι ανηλίκοι που αποτελεί πρόκληση για τις διοκτικές αρχές. Επίσης, ε, ο εξαναγκασμός και ο εκβιασμός ε, αποτελεί μια αυξανόμενη απειλή για την κοινωνία μας και τέλος εδώ πέρα θα ήθελα να αναφέρω το ότι αυξάνεται η κακοποίηση εξ με streaming, με ζωντανή μετάδοση. Τέλος, στο σκοτεινό δίκτυο, έχουμε μια αύξηση μεμονωμένων μαγαζιών και όχι πλέον site που προσφέρουν τα πάντα, αλλά πιο εξειδικευμένα. Όπως είπαμε, είναι ένα περιβάλλον με κινητικότητα Και βλέπουμε ότι αυξάνονται και οι διάφορες πλατφόρμες μηνυμάτων. Επόμενη διαφάνεια. Τι κάνει η Europol λοιπόν με την έκθεση αυτή προς τα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να το αναφέρω και αυτό, γιατί αναφέρουμε όχι μόνο τις απειλές αλλά και τα αποτελέσματα. Η Europol δημιούργησε μια συγκεκριμένη ομάδα για το σκοτεινό δίκτυο και στα αριστερά βλέπετε το τι κάναμε, κάποια site που κατεβάσαμε σε συνεργασία με κάποια κράτη-μέλη. Δεύτερον έχουμε το Power Off σε συνεργασία με τις διοκτικές αρχές για να κατεβάσουμε το οργάνωση Web Stressor που προσέφερε κατά παραγγελία επιθέσεις ε, την άλλο Service. Ε, υπήρχαν χιλιάδες πελάτες αυτής της υπηρεσίας που πλήρωναν ε, μία μήνυα συνδρομή και για 15 ευρώ το μήνα μπορούσε κανείς να παραγγείλει μία επίθεση. Κατεβάσαμε λοιπόν το site αυτό, το οποίο οδήγησε σε πολλές έρευνες όχι μόνο των προμηθευτών αλλά και όσων έκαναν τις παραγγελίες. Ένα τρίτο παράδειγμα που θα ήθελα να αναφέρω αφορά τη σεξουαλική κακοποίηση. Μια έρευνα που ξεκίνησε το 2019 στα κράτη-μέλη με βάση πληροφορίες μας έδωσε η και οι Αμερικανοί ομολόγοι μας και καταλήξαμε στην ταυτοποίηση ενός ατόμου που δούλευε σε μια χώρα και ζούσε σε μια άλλη και με συντονισμένη δράση ε, ερευνήθηκε το σπίτι του και χρησιμοποιούσε πάνω από 40 διαφορετικά προφίλ στο διαδίκτυο σε διάφορες πλατφόρμες για να προσεγγίζει θύματα και είχε διάφορους λογαριασμούς για μηνύματα, για να κανονίζει και με άλλους ενηλίκους να κακοποιήσουν το ίδιο παιδί. Οπότε αυτοποιήθηκαν όλοι οι ύποπτοι και τα παιδιά και η έρευνα συνεχίζεται. Και για να διδαχτούμε από τέτοιες έρευνες επίσης προσπαθούμε να στήσουμε νέες δραστηριότητες όπως η εβδομάδα ηλεκτρονικής περιπόλου όπου προσκαλούμε κράτη-μέλη στο αρχηγείο μας για να δούμε ακριβώς ε, το τι γίνεται ε, για να μάθουμε και όλες να δαχτούμε ένας από τον άλλον για να υπάρχουν ε, για να δούμε τις δραστηριότητες που υπάρχουν στις σκοτεινές αγορές. Επόμενη διαφάνεια. Συστάσεις. Τις βλέπετε εδώ πέρα. Θα τις αναφέρω. Κατά την απόψή μας απαιτείται μια διεθνός συντονισμένη προσέγγιση και επίσης να ξέρουμε τι κάνουμε ο καθένας επιχειρησιακά, δεδομένου του ρόλου πλέον του εγκλήματος ως υπηρεσία θα πρέπει να στοχεύσουμε τους παρόχους, γιατί θα είμαστε πιο επιτυχείς. Επίσης χρειάζεται μια διεπιστημονική προσέγγιση για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια στο διαδίκτυο και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δούμε και τις εκστρατείες εκπαίδευσης. Επίσης, πρέπει να συνεισφέρουμε στην κυβερνοεκπαίδευση και ανθεκτικότητα. Αυτό το κάνουμε και για όσους ε, μεταφέρουν χρήματα και για τους εκβιαστές και πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα θα πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να ενισχύσουμε περαιτέρω αυτήν την συνεργασία, γιατί αυτοί έχουν τις βασικές πληροφορίες που χρειαζόμαστε. Και έτσι νομίζω ότι η συνεργασία αυτή πρέπει να αποτελέσει μια καινοτομία, να έχουμε νέους τρόπους εργασίας και μια πιο γρήγορη προσέγγιση στον τομέα αυτών. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα στην επόμενη διαφάνεια προσπαθούμε να βρούμε και νέους τρόπους να διαταράξουμε το επιχειρησιακό τους μοντέλο. Απλά τονίζω μία δραστηριότητα εδώ που κάνουμε εδώ και τρία χρόνια, το site όχι άλλα λίτρα, καθώς τα άλλη τρισμικά αυξάνονται για να δούμε πώς θα διαταράξουμε το μοντέλο των εγκληματιών, έτσι ώστε να μην είναι πλέον δυνατόν να αποσπάσουν χρήματα. Συμφωνήσαμε λοιπόν με δύο ιδιώτες εταίρους και άλλες διοκτικές αρχές να στήσουμε αυτό το site και κάθε, εταιρεία, συμφωνήσαμε, θα ε, είχε ε, εργαλεία αποκρυπτογράφησης ε, στο site αυτό και το προσφέρουμε δωρεάν σε όλους τους πολίτες της Ευρώπης και παραπέρα. Ξεκίνησα με τέσσερις εταίρους, αλλά βλέπετε εδώ πέρα πώς Τελικά έχουμε πάνω από 150 συνεργάτες ε, από διάφορους ε, κλάδους, ε, από αυτούς που δίνουν δωρεάν τα εργαλεία από κρυπτογράψεις, έτσι σπάμε το επιχειρηματικό τους μοντέλο και βλέπετε τα αποτελέσματα για το τι αποτελέσματα έχουμε. Δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό το site, γίνεται παγκόσμιο πλέον. Η συνεργασία αυτή σημαίνει ότι είναι επίσης ε, διαθέσιμο σε 36 γλώσσες. Χρησιμοποιείται ανά τον κόσμο. Βλέπετε εδώ πέρα ότι ο αριθμός των θυμάτων ε, και έχουμε κάνει εδώ μια πολύ προσεκτική εκτίμηση είναι πάνω από 200.000 άνθρωποι υπολογίζουμε τον αριθμό των λίτρων σε πάνω από 100 εκατομμύρια που δεν ε, πληρώθηκαν ε, σε πάνω από 188 χώρες. Και βεβαίως αυτό είναι υποφελές για όλους γιατί διαταράσσουμε ε, το μοντέλο των εγκληματιών και βεβαίως οι εταιρείε τα δίνουν όλα δωρεάν αλλά μετά βεβαίω θα φροντίσει να εξασφαλιστείς για το μέλλον, οπότε και κερδίζουν και οι εταιρείε. Ένα άλλο παράδειγμα που θα ήθελα να σας αναφέρω αφορά τη σεξουαλική κακοποίηση. Ένα site ε, το οποίο στήσαμε πριν από δύο χρόνια για να βοηθήσουμε τις ε, διοκτικές αρχές να κάνουν έρευνες ε, που έχουν ε, κολλήσει κάπως ε, στα θέματα αυτά και να βρούμε νέες πληροφορίες. Και το σκεπτικό ήταν να χρησιμοποιήσουμε εικόνες σχετικές και να ζητήσουμε από το κοινό να μας βοηθήσει να ταυτοποιήσουμε αυτά τα αντικείμενα. Δηλαδή, αντί να αναζητούμε κάτι σε 200 χώρες, ε, αν έχουμε μια φωτογραφία και κάτι φαίνεται στο φόντο, μπορούμε να το περιορίσουμε σε 10-20 χώρες. Και αυτό θα το έβλεπε είτε το κοινό είτε η ειδική. Αυτό για τις περιπτώσεις οι οποίες είχαν καταλήξει σε αδιέξοδο λόγω έλλειψης πληροφοριών. Ξεκινήσαμε λοιπόν με τη δημοσίευση 20 εικόνων. Ε, ξεκινάω με αυτήν εδώ. Ε, κάντε λίγο πίσω. Λοιπόν, εδώ βλέπετε. Ξεκινήσαμε με 20 μηνύμα εικόνες τις πρώτες εβδομάδες λάβαμε 4.000 email από ανθρώπους που ήθελαν να μας βοηθήσουν και οι εικόνες που δημοσιεύονται τώρα είναι 190 σχεδόν και λάβαμε 24.000 πληροφορίες από το κοινό για να μας βοηθήσει να, να γνωρίσουμε αυτά τα αντικείμενα. Δεν θεωρούσαμε επίσης ποτέ ότι θα λύναμε ποτέ ε, τα εγκλήματα, αλλά ε, εννέα παιδιά ταυτοποιήθηκαν και δύο εγκληματίες ε, έχουν διωχθεί. Βλέπετε εδώ πέρα τι δημοσιεύουμε ακριβώ. Βλέπετε παραδείγματος χάρη ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. και δημοσιεύσαμε ακριβώς, βρήκαμε ακριβώς που ήταν το ξενοδοχείο. Να, αυτό εδώ. Εδώ πέρα βλέπετε μια μπανιέρα. Το βάλαμε Παρασκευή βράδυ στο διαδίκτυο και λίγα λεπτά αργότερα το βράδυ μας έστειλαν την εικόνα που βλέπετε στα δεξιά και το ταυτοποιήσαμε. Οπότε το κοινό, το πλήθος μας βοηθάει να βρούμε πού βρίσκονται διάφορα μέρη και να ξεκινήσουν έτσι οι έρευνες Τότε με αυτόν τον τρόπο βλέπετε πώς ε, μπορούμε να βοηθηθούμε. Βλέπετε επίσης ε, ε, τον τύπο που έγραψε γι' αυτό. Επόμενη διαφάνεια για το μέλλον. Ποιες είναι οι εξελίξεις που βλέπουμε. Τα λιτρισμικά θα παραμείνουν στην πρώτη θέση. Θα υπάρχουν πιο εξειδικευμένοι πάροχοι εγκλήματος ως ε, υπηρεσία και νομίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα μια αγορά η οποία αυξάνεται. Αναμένουμε να δούμε επίσης αύξηση στις επιθέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα θα είναι επιτυχής ε, γιατί οι εταιρείε ε, συνεχώς ε, αναθέτουν κομμάτι της λειτουργίας τους σε άλλες εταιρείε. Το λεγόμενο phishing επίσης θα συνεχίσει να παραμένει σημαντικό με πιο εξειδικευμένους και επαγγελματικούς τρόπους προσέγγισης ανθρώπων που έχουν ρόλο κλειδί σε μια εταιρεία. Ανέφερα ήδη τα νέα συστήματα πληρωμών που προκύπτουν και τα χρησιμοποιούν οι εγκληματίες αλλά και επιτίθενται σε αυτά και η τεχνολογία deepfake ε, επίσης ε, θα αυξηθεί. Συμπερασματικά λοιπόν, τι ε, πρέπει να γίνει ως αντίδραση από τις διοκτικές αρχές. Γνωρίζω ότι υπάρχει μια πρόταση της ε, Κομισιόν για ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία. Στις περισσότερες έρευνες, 85% τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία είναι κομμάτι της δραστηριότητας και θα συνεχιστεί αυτό. Και επίσης το σύστημα βίας νομικής αρρωγής που έχουμε τώρα είναι μάλλον θα έλεγα ξεπερασμένο. Χρειάζεται πολύς χρόνος και ο χρόνος ε, δεν περισσεύει ε, όταν μιλάμε για το διαδίκτυο οπότε πρέπει να υπάρχει άμεση συνεργασία με αυτούς που έχουν τις ε, πληροφορίες ναι, για να υπάρχει εποπτεία. Βεβαίω, γνωρίζω πως βεβαίως η Λίμπε συζητά αυτά Υπάρχει ήδη δημοσιευτεί ένα πρώτο σχέδιο και κάποιες ιδέες δικές μας και ανησυχίες που αφορούν το θέμα επίσης. Ειδικά επίσης για το πώς θα μπορέσουμε να δούμε από πού ξεκινάει το έγκλημα, διευθύνσεις δηλαδή διαδικτύου. Υπάρχουν αυστηρές ε, διατάξεις για αυτή την πολύ βασική πληροφορία. Είναι μια πληροφορία όμως που απαιτείται και δεν θα πρέπει να περιορίζεται αυτό σε μερικά μόνο εγκλήματα το κατόφλι για τα ευαίσθητα δεδομένα. Υπάρχει μια πρωτοσύνη να ανέβει από τα 3 στα 5 χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι και δύσκολο για να υπάρχει και αυτή η ανταλλαγή εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης γιατί σε κάποιες χώρες δεν τιμωρείται αρκετά αυτό. Οπότε ζητάμε να δείτε ακριβώς τον αριθμό των ετών που απαιτείται ως κατοφλή και τέλος ε, επανέλθω στην δικαστική συνεργασία ως αρχή. Είναι μια αρχή η οποία θα πρέπει να παραμείνει αλλά ταυτόχρονα υπάρχει ανάγκη να μην έχουν τόσα εμπόδια διοκτικές αρχές. Νομίζω λοιπόν ότι απαιτείται οι διοκτικές αρχές να έχουν τα εργαλεία αυτά να μπορούν να διατηρήσουν τα δεδομένα, η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και η πρόσβαση σε βάσεις ε, δεδομένων. Αυτά κοιτάμε και ευχαριστώ να τα συζητήσουμε μαζί σας. Σας ευχαριστούμε κύριε Φανκέμερτ. Έχω δει ότι ήδη κάποιοι συνάδελφοι ζήτησαν το λόγο. Παρακαλώ ε, σηκώστε τώρα είτε το χέρι σας είτε το καρτελάκι σας για να συμπληρώσουμε τον κατάλογο μιλητών. Και ξεκινάμε με την κυρία Σίπελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να εκφράσω κυρίως κάποια ερωτήματα. Και πάλι συζητάμε το ζήτημα της κρυπτογράφησης και το πρόβλημα που η κρυπτογράφηση δημιουργεί στις προσπάθειες των διοκτικών αρχών να ακολουθήσουν την επικοινωνία των εγκληματιών. Ωστόσο, δεν, δεν θα συμφωνήσετε ότι εάν αυξηθεί ο αριθμός των φυσικών και νομικών προσώπων που χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση, ε, αυτό θα βοηθήσει έτσι ώστε να αντισταθούμε σε όλες αυτές τις απειλές όλο και περισσότερο. Το δεύτερο, όλο και πιο συχνά μιλούμε για κυβερνοεπιθέσεις. Πιστεύετε ότι συνεχίζει να υφίσταται ένα πρόβλημα με την υποδομή ή ε, με μια ε, κατάσταση στην οποία δεν γνωρίζουν όλοι πώ να δημιουργήσουν ένα ασφαλέ περιβάλλον. Είτε πρόκειται για μια επιχείρηση, είτε πρόκειται για άλλου τομεί. Δηλαδή δεν υπάρχει εμπιστητοποίηση. Τρίτον, μιλήσατε ήδη για την αύξηση του υλικού από, τους, από τα ίδια τα παιδιά που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σεξουαλική εκμετάλλευση, κακοποίηση για πολλούς και διάφορους λόγους και είπατε ότι αυτή η τις συστάσεις του φαινομένου δεν μπορεί να έρθει μόνο από την αστυνομία αλλά επίσης χρειάζεται και ευαισθητοποίηση και πιθανώς μια συνεργασία και με τα σχολεία. Είναι μια από τις συστάσεις σας. Λοιπόν, το ερώτημά μου είναι το εξή. Βλέπετε να έχουν υπάρξει εξελίξεις στον τομέα αυτό στα κράτη-μέλη, πρωτοβουλίες δηλαδή για την ε, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση των παιδιών, έχει αρχίσει να συζητιέται το θέμα. Στο τέλος επίσης της παρουσίασής σας μιλήσατε και για αυτή τη διαδικασία με την οποία προσπαθείτε να ταυτοποιήσετε αντικείμενα στο φόντο ε, μιας ε, φωτογραφίας και πόσο χρήσιμο είναι το να απευθύνεστε στο κοινό για αυτό. Όμως το ερώτημα μου είναι το εξής δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τις συστήματα αντίστροφης αναζήτησης εικόνων στο ίντερνετ για να ταυτοποιήσετε με αυτόν τον τρόπο την τοποθεσία. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Κύριε Ρίκμοντ. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Έχω μερικές ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα για την τεχνολογία deepfake. Μιλήσατε ήδη για αυτήν και με αυτό, βάσει αυτό που διαβάζω στην έκθεση, οι εξελίξεις στον τομέα αυτό του deepfake, δηλαδή την δημιουργία μιας ε, ψεύτικης εικόνας με τη χρήση των βαθία της βαθίας μάθησης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για, είτε για τη δημιουργία φωτογραφιών σεξουαλικής ε, κακοποίησης, είτε και για την ταυτοποίηση των δραστών. Θα ήθελα να μου πείτε αν έχετε αξιοποιήσει αυτή την τεχνολογία για την ε, ταυτοποίηση των θυμάτων και ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις που έχετε αντιμετωπίσει. Μετά. Για το ζήτημα του εικονικού βιασμού. Πού βρισκόμαστε και θεωρείτε ε, ότι μπορεί η κακοποίηση ενός παιδιού να, θεω... διωχθεί στο πλαίσιο ενός... Ε, στο ίδιο πλαίσιο λοιπόν. Τρίτο ερώτημα. Βλέπουμε ότι τα κοινωνικά μέσα δικτύες χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για την διευκόλυνση του κυβερνού Πώς, Πώ πιστεύετε ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε την ενημέρωση του κοινού. Φαίνεται επίσης ότι η καταπολέμηση των, των πηγών χρηματοδότησης, περιορισμός τους είναι πολύ σημαντικός. Αυτό που κάνουμε επαρκεί προς αυτή την κατεύθυνση. Γνωρίζω επίσης ότι υπάρχει και η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού στις αστυνομικές αρχές, στα διάφορα κράτη-μέλη που χρειάζεται για να συνεχίσουν μια δίωξη. Έχουμε όλο και περισσότερα εργαλεία, όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε τη σημασία του ανθρώπινου δυναμικού. Τι κάνει λοιπόν η Europol για να βοηθήσει τα κράτη-μέλη στο επίπεδο αυτό. Και τελευταία μου ερώτηση. Μία από τις ε, συστάσεις της έκθεσης για να αντιμετωπιστούν και οι φυστάμενες αλλά και πιθανές μελλοντικέ απειλές είναι να δημιουργηθεί ένας κόμβος, hub, για την συνεργασία των ε, πιο ε, σημαντικών διοκτικών αρχών και άλλων αρχών που έχουν σχέση με το θέμα. Μπορείτε να μας δώσετε λίγο περισσότερες πληροφορίες, λίγο μεγαλύτερη λεπτομέρεια σε σχέση με την πρότασή σας αυτή και πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσε να υλοποιηθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κέρνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και για αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση, τον προσκεκλημένο μας. Ευχαριστώ. Να σας συγχαρώ για την ιδέα για την ε, αξιοποίηση των πληροφοριών από το κοινό για την ταυτοποίηση των διαφόρων αντικειμένων στο φόντο μιας φωτογραφίας. Ε, θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς το δημοσιοποιείτε αυτό, πώς φροντίζετε να είναι γνωστό στο, στο κοινό, στον κόσμο για να γνωρίζει ότι μπορεί να βοηθήσει με αυτόν τον τρόπο έτσι ώστε να την δει τη φωτογραφία σου το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων. Μετά αναφερθήκατε στη σημασία των πιστηρίων και αν κατάλαβα καλά. Είπατε ότι το βασικό είναι να μπορείτε να ταυτοποιήσετε ποιο πρόσωπο χρησιμοποίησε μια διεύθυνση IP. Αυτό ε, το ονομάζουμε δεδομένα πρόσβασης. Οι ανάγκες σας λοιπόν εστιάζονται περισσότερο στα δεδομένα πρόσβασης, να μπορείτε να ταυτοποιήσετε ποιος βρίσκεται πίσω από μια διεύθυνση IP και θα μπορούσε να σας διευκολύνει δηλαδή μια πρόσβαση σε αυτό το στοιχείο, ενώ κατά τα άλλα για άλλα δεδομένα τα οποία μπορεί να είναι περισσότερο ευαίσθητα και να θέτουν ζητήματα θεμελιωδών ελευθεριών, οι ασφαλιστικές δικλείδες να είναι πιο αυστηρές. Γιατί Ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στι ανάγκε των διοκτικών αρχών και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Επομένω, θα ήθελα να μου πείτε, εσεί αν είχατε πρόσβαση στα δεδομένα πρόσβαση, αυτό θα επαρκούσε έτσι ώστε να κρατήσουμε πιο αυστηρέ ε, διαφορετικέ ασφαλιστικέ δικλείδε και διαφορετικά μέσα πιθανώ για την πρόσβαση σε άλλα δεδομένα που μπορούν να είναι πιο ευαίσθητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Ντυπό. Ευχαριστώ και εγώ για την έκθεση και την εικόνα που μας δώσατε. Ο ερώτημά μου πηγαίνει προς παρόμοια κατεύθυνση με αυτό της κυρίας Κέρνερ. Είδα πως είστε πολύ δραστήριοι στο Instagram. Όχι μόνο για την κακοποίηση παιδιών, αλλά και για άλλα ζητήματα που προσπαθείτε να ζήσετε μέσω του κοινού. Μπορούσε να μεταφερθεί και σε άλλους ε, τομείς και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλύτερα για να ε, εμποδίσουμε τέτοια εγκλήματα. Σας ευχαριστώ. Κυρία Κέλλαρ. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να μιλήσω στα γαλλικά. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση της έκθεσης ε, της αξιολόγησης απειλών. Ε, πραγματικά είμαστε ευγνώμονες για το αξιοθαύμαστο σα έργο, ιδιαίτερα στα θέματα παιδική πορνογραφία και σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών. Είναι σημαντικό να προστατεύσουμε τα παιδιά μα από σεξουαλική εκμετάλλευση κάθε είδους. Φάνηκε η ευγνωμοσύνη μα και από τι παρεμβάσει των συναδέλφων. μπορείτε να μα περιγράψετε πώ συνεργάζεστε με του εθνικού φορεί, γιατί η διαφάνεια για τους εταίρους δεν ήταν πολύ σαφής είδα ότι η γαλλική αστυνομία ήταν ε, ε, πολύ χαμηλά στον κατάλογο των συνεργατών. Πώς ε, συνεργάζεται λοιπόν με εθνικούς ή άλλους ειδικευμένους φορείς. Δεύτερη ερώτηση. Μιλούμε όλο και περισσότερο για την κατάσταση των μεταναστών. Οι οικογένειες μεταναστών είναι θύματα εκμετάλλευσης για να πληρώσουν και τους λαθροδιακινητές ε, ε, από τις χώρες προέλευση αλλά και για τη διέλευσή τους στην Αφρική όταν έχουν στόχο να έρθουν στην Ευρώπη. Χρειάζονται χρήματα σε όλη τη φάση της, ε, του ταξιδιού τους ε, όταν εξαρτάται η επιβίωση τους από τους λαθροδιακινητέ και οι οικογένειές του γίνονται θύματα εκμετάλλευση για να βρεθούν αυτά τα χρήματα. Πώς θα αποτρέψουμε αυτή την αύξηση της επιρροή των λαθροδιακινητών και τη ικανότητα τους να εκβιάζουν τις οικογένειες και να τους ε, παίρνουν χρήματα για να εξασφαλίσουν την επιβίωση των μεταναστών. Ο κύριος Μάντισον. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα μιλήσω Νικά. Ε, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε, Είδα τα στατιστικά στοιχεία για τους ανηλικούς στην Εστονία. Το ερώτημά μου είναι ποιες χώρες συνεργάζονται περισσότερο όταν μιλάμε για πλατφόρμες ε, του διαδικτύου που χρησιμοποιούνται για εγκλήματα κατά ανηλίκων. Και τι έχει κάνει η Europol για να διαλευκάνει τέτοια εγκλήματα. Έχετε δεδομένα και αναλύσεις για το πόσοι από τους ε, δράστες ε, που πιάσατε είναι υπότροποι και πόσοι ε, το έκαναν για πρώτη φορά. Επίση είναι διαφορετική εγκληματικότητα στα κράτη-μέλη Και βεβαίως αυτά τα πράγματα επηρεάζουν κάποιον μια ολόκληρη ζωή. Οι ποινέ όμως, άμα δεν περιλαμβάνουν φυλάκιση, είναι πολύ ήπιε. Και αναφέρθηκε επίσης το θέμα της μετανάστευση. Πριν από κάτι χρόνια η Ευρώπη σοκαρίστηκε για το ότι είχαμε μαζικά περιστατικά σε γερμανικές πόλεις όπου είχαμε ε, εκμετάλλευση γυναικών από μετανάστες και τέτοια. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου έχει υπάρξει σεξουαλική κακοποίηση παιδιών από μετανάστες. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μιλήσατε για τον διεθνή συντονισμό και τη βελτίωση που πρέπει να επέλθει. Θα ήθελα να μας δώσετε κάποια παραδείγματα για το πού κατά την άποψή σας πρέπει να δράσουμε γρηγορότερα. Χτες είχαμε επίσης την πρώτη κοινή συζήτηση για τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία και διαπίστωσα πως το θέμα αυτό κινδυνεύει να εξασθενήσει και να μην είναι καθόλου αποτελεσματικό τελικά. Γι' αυτό το ερώτημά μου είναι το εξής. Ε, Φενός αν μπορείτε να δείτε τα θεμελιώδη δικαιώματα από την, άλλου, από την άλλη βεβαίως ε, της ε, διαδικασίας. Γιατί πρέπει βεβαίως να εκπληρώνει και τον σκοπό του ο κανονισμός, έτσι. Σας ευχαριστώ. Κυρία αλσα αλ Καταπληκτικά δηλαδή, προφέρατε το όνομά μου, κύριε Πρόεδρε. Μπράβο σας. Θα μιλήσω σου ειδικά όμως. Ευχαριστώ για αυτή την πολύ σημαντική και διαφωτιστική παρουσίαση. Καλά δεν είπα ότι θα μιλήσω σου ειδικά. Εν πάση στα σου ειδικά. Έχω δύο ερωτήσεις προς το Διευθυντή των Επιχειρήσεων της Ευρωπόλ. Η πρώτη ερώτηση αφορά την αξιολόγηση που κάνετε εσείς για την κατάσταση. Στις σκανδιναβικές χώρες, πολλής λόγος γίνεται για ένα ευρωπαϊκό FBI. Ποια είναι η άποψή σας? Πιστεύετε ότι ένα ευρωπαϊκό FBI θα οδηγήσει στη διαλεύκανση περισσότερων υποθέσεων? Ή αρκεί η συνεργασία για την εξυχνίαση τέτοιων εγκλημάτων, πιστεύετε. Δεύτερη ερώτηση. Τι κατά τη γνώμη σας εμποδίζει την επιτυχία της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας. Πού έγινε τα προβλήματα, δεν έχουμε αρκετούς μηχανισμούς, δεν υπάρχει αρκετή εναρμόνιση, υπάρχει απροθυμία από τους εθνικούς φορείς για την ανταλλαγή πληροφοριών. Είναι κάτι δηλαδή που επαφείται ή που, κάτι για το οποίο ευθύνονται οι αρχές που επιλαμβάνονται αυτών των θεμάτων. Ο κύριος Κόφωτ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον αναπληρωτή εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπόλ για την παρουσίασή του. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι γίνεται με τις ειδικέ δανέζικες ρυθμίσεις συνεργασίας με την Ευρωπόλ. Ξέρω ότι ε, ισχύουν ειδικέ διατάξεις για τη Δανία στα θέματα αυτά. Μπορείτε να μας ενημερώσετε για την δανέζικη συμμετοχή στη συνεργασία, αυτή την αστυνομική συνεργασία. Μακάρι να πείτε ότι είναι εξαιρετική συνεργασία μεταξύ της Ευρωπόλ και της Δανικής Αστυνομίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ε, όσοι ζήτησαν το λόγο τον έλαβαν. Δεν βλέπω άλλο κανένα να θέλει να μιλήσει, οπότε επανέρχομαι στους καλεσμένους μας. Ο κύριος Βαχέμερτ θα λάβει και πάλι το λόγο για να απαντήσει. Έχει χρόνο μέχρι τις 10:30 και μισή, ένα τέταρτο, δηλαδή για να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις που του υποβλήθηκαν. Ευχαριστώ, θα κάνω την μπορώ κύριε Πρόεδρε. Και τις πιο ειδικές ερωτήσεις θα τις παραπέμψω στον συνάδελφο τον Φερνάντο για την κρυπτογράφηση ως σύστημα. Και εμείς ως ε, διεκτική αρχή θεωρούμε ότι είναι πολλά τα ωφέλη της κρυπτογράφησης και κάνει την ε, κοινωνία μας την εικονική πιο ασφαλής. Βέβαια, αν γίνεται κατάχρηση της κρυπτογράφησης από εγκληματίες, θα πρέπει να μπορούν οι διεκτικές αρχές ε, στο νομικό πλαίσιο να έχουν πρόσβαση σε αποκρυπτογράφηση. Οπότε θέλουμε ε, να αναπτύξουμε αισθήματα, όπως κάναμε και με τις υποκλοπές. Να προβλέψουμε τις νομικές διατάξεις για να αφαιρέσουμε την κρυπτογράφηση για να περιφρουρήσουμε και τα δικαιώματα των θυμάτων. Σε ό,τι αφορά την ευαισθητοποίηση του κοινού για την παιδική πορνογραφία και την σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών, βοηθούμε τα κράτη-μέλη και συμμετέχουμε στην οργάνωση ε, εκστρατιών ευαισθητοποίησης που χρησιμοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι σε μερικές χώρες μόνο. Και μάλιστα αυτή τη εβδομάδα είχαμε μια εκστρατεία στη Βουλγαρία που είχε μεγάλη επιτυχία. Προσπαθούμε λοιπόν όχι μόνο να συνεργαζόμαστε σε θέματα ε, διερεύνησης υποθέσεων, αλλά και στην διοργάνωση εκστρατιών ευαισθητοποίησης. Σε ό,τι αφορά το outsourcing, έχουμε ε, χρήση της τεχνολογίας έτσι. Βέβαια, οι διεκτικές αρχές ε, περιορίζονται στις δικές τους δραστηριότητες και το crowdsourcing μας βοηθάει μερικές φορές, αλλά σε δεδομένα όρια και πλαίσιο. Έχουμε και εταιρείε όπως το Reddit, όχι μόνο το κοινό που μας βοηθούν ε, και στον εντοπισμό των του τόπου χάρη στο φόντο αυτών των ε, φωτογραφιών, των εικόνων. Και μας έχει βοηθήσει και το crowdsourcing, η συμμετοχή του κοινού και οι πληροφορίες που λαμβάνουμε από αυτούς για την ταυτοποίηση κάποιων χώρων. Το θέμα της τεχνολογίας deepfake θα το αφήσω για τον Φερνάντο. Σε ό,τι φορά τις ομάδες, τι τρομοκρατικέ, με την αρμόδια ομάδα ε, έχουμε κατεβάσει παράνομο περιεχόμενο και έχουμε επισημάνει το ζήτημα στις αρμόδιες, στις υπεύθυνες ε, εταιρείες που παρέχουν τις υπηρεσίες. Έχουμε παραπέμψει πάνω από χίλιες σελίδες οι λογαριασμούς Twitter από τις εταιρείες αυτές. Και μάλιστα μέχρι 90% του περιεχομένου που παραπέμπουμε τελικά κατεβαίνει. σε περίπτωση που υπάρχει παράνομο περιεχόμενο, γίνεται αυτή η παραπομπή προκειμένου να αφαιρεθεί. Τώρα, η χρήση του Ιντερνετ για τη ριζοσπαστικοποίηση. Το πρόβλημα είναι ότι μερικέ φορέ δεν ε, γίνεται αυτή η απόπειρα σε ανοιχτό Ιντερνετ, αλλά σε ειδικού διάβλου επικοινωνία, στους οποίες δεν έχουμε πρόσβαση. Προσπαθούμε πάντω να εντοπίσουμε και νέε μεθόδου για τη χρήση των μέσων κοινωνική δικτύωση και να καταλάβουμε καλύτερα το πώς χρησιμοποιούνται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε κάθε επίθεση πάντως ε, ο ρόλος μας είναι να εντοπίσουμε πώς οι δράστες της επίθεσης ε, είναι παρόντες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και προσπαθούμε σε συνεργασία με τις διοκτικές αρχές να εκκινήσουμε τις έρευνες. Τι γίνεται με την ευαισθητοποίηση, ε, με ρώτησε κάποιο. Έχουμε ειδικέ εκστρατείε. Πρόσφατα είχαμε την εκστρατεία ε, «Το έγκλημα δεν γνωρίζει φίλο, δεν έχει φίλο». Επίσης, προσπαθούμε να εγείρουμε την ευαισθητοποίηση για τις εγκληματικέ δραστηριότητες γενικώ. Και γι' αυτό έχουμε τις ιστοσελίδες μας που έχουν πολλές επισκέψεις, από 8 μέχρι 200.000 τη μέρα επισκέψεις, ειδικά, ειδικά όταν έχουμε κάποιε εκστρατείε. Και μάλιστα σε δύο εβδομάδε είχαμε πέντε συλλήψει. ε, κάτι που δείχνει πόσο χρήσιμο είναι αυτό το crowdsourcing, χρήση των πληροφοριών από το κοινό. Μερικέ φορέ εγγύρουμε την ευαισθητοποίηση προσφέροντα τι υπηρεσίε μα και στι ευρωπαϊκέ διεκτικέ αρχές. Σε ό,τι αφορά τι ηλεκτρονικέ ε, αποδείξει, τα αποδεικτικά στοιχεία, ε, φυσικά η πρόσβαση είναι ένα θέμα, αλλά δεν είναι το μόνο και τα μεταδεδομένα έχουν μεγάλη σημασία στην ε, έρευνα. Οπότε, σε μία ε, νομική έρευνα καλό θα ήταν να υπάρχει δυνατότητα πρόσβαση σε τις πληροφορίες για τις πιο ε, σοβαρές υποθέσεις. Εκεί υπάρχει ένα όριο, ένα κατόφλι στην ανταλλαγή δεδομένων και όταν είναι πολύ ψηλό το κατόφλι χάνουμε πολλές πολύτιμες πληροφορίες ε, και ίσως η πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές θα μας επέτρεπε να προστατεύσουμε καλύτερα τα θύματα. Και ούτως ή άλλως ο δικαστής είναι ο τελικός επόπτης αυτής της διαδικασίας, οπότε χρειάζεται και πρόσβαση αλλά και μεταδεδομένα. Η πλατφόρμα που χρησιμοποιούμε. Ο ρόλος της Ευρωπόλ είναι μια, ένας ρόλος πλατφόρμας και ακριβώς ε, επειδή είμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και διοργανώνουμε τις εξτρατείες πανευρωπαϊκά έχουμε ένα καλύτερο εποπτικό ρόλο. Και είμαστε ο σύνδεσμος μεταξύ αυτών που θέλουν οι υπηρεσίες με αυτούς που τις προσφέρουν. Αυτό είναι ο ρόλος της Ευρωπόλ για τις διοκτικές αρχές. Έχουμε αυτό το συνδετικό ρόλο δηλαδή. Συνεργασία με εθνικούς φορείς. Συνεργαζόμαστε και με όλα τα κρατημέλη αλλά και με τρίτους εταίρους με τους οποίους έχουμε συνεργασ... συμφωνίες συνεργασίας και γίνεται τακτική ενημέρωση για το βαθμό συνεργασίας. Και μάλιστα στον κανονισμό μας υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης ε, που θα υποβάλλουμε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το βαθμό συνεργασίας που έχουν τα κράτη-μέλη με την Ευρωπόλ. Εκμετάλλευση των μεταναστών. Το βλέπουμε αυτό. Ιδιαίτερα στις των μεταναστών και στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Εκεί έχουμε πολύ ε, αμήλικτη παρέμβαση και το οργανωμένο εγκλήματος. Είχαμε πρόσφατα το θάνατο περίπου 40 μεταναστών στο ψυγείο που βρέθηκαν. Και προσπαθούμε να βρούμε τους τρόπους λειτουργίας ε, και τη μεθοδολογία των σπυρών, χρησιμοποιώντας και τις τεχνολογίες και όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Τώρα, αν χρεια... ως προς την ερώτηση για το αν χρειαζόμαστε ε, βελτίωση της διεθνούς συνεργασίας. Όντως, το δικό μας σύστημα ε, στηρίζεται στα δικαιοδοτικά, όρια. Ενώ το κυβέρνο έγκλημα δεν γνωρίζει σύνορα, δεν γνωρίζει όρια. Οπότε η δικαστική συνεργασία είναι μερική απόκριση στις ανάγκες μας. Και πολλές πληροφορίες που έχουμε για το έγκλημα δεν βρίσκονται στα χέρια μιας κυβέρνησης ή κυβερνητικών φορέων, αλλά στα χέρια ιδιωτών εταίρων. Και γι' αυτό είναι σημαντική η συνεργασία και η νόμιμη πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές υπό τον έλεγχο των δικαστήριων. Και τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία έχουν μεγάλη σημασία. Θα πρέπει λοιπόν η πρόσβαση σε αυτά να γίνεται στα πλαίσια και του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Θα πρέπει να υιοθετήσουμε μια αποτελεσματική προσέγγιση λοιπόν και στα θέματα αυτά. Τώρα, χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό FBI, ρώτησε μια κυρία από τη Σουηδία. Αυτό δεν είναι ένα θεσμικό ερώτημα που καλούμαστε εμείς ως Ευρωπόλ να απαντήσουμε. Η ανάγκη για ένα ευρωπαϊκό FBI προϋποθέτει ένα ομοσπονδιακό σύστημα. Δεν έχουμε όμως τέτοιο ομοσπονδιακό νόμο. Εγώ θεωρώ ότι δεν χρειαζόμαστε τόσο ένα ευρωπαϊκό FBI, αλλά μια ευρωπαϊκή αστυνόμευση για να κάνουμε τα πράγματα με το δικό μας τρόπο, τον ευρωπαϊκό. Και η Ευρωπόλος πλατφόρμα προσπαθεί να διευκολύνει τις διοκτικές αρχές να ασκήσουν καλύτερα το ρόλο, της, το ρόλο τους. Και επίσης να αναβαθμίσουμε και τη γνώση των εμπειρογνωμόνων στα κράτη-μέλη. Με την Task Force για το ταυτοποίηση θυμάτων. Εκεί συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη και στη δικά μας γραφεία και προσπαθούμε να επιτύχουμε ένα διπλό αποτέλεσμα. Πρώτα να το, ε, εντοπίσουμε τους δράστες και να ε, βελτιώσουμε την επιμόρφωση των ε, εμπειρογνωμόνων. Και φυσικά η πρόληψη είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Και φυσικά αν παραμείνουμε στα παραδοσιακά και συστήματα δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε αποτελεσματικές λύσεις στα προβλήματα. Σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις με τη Δανία, έχουμε στενή συνεργασία και ειδικέ ρυθμίσεις για την συνεργασία με τη Δανία. Η Δανία δεν έχει άμεση πρόσβαση σε όλες τις βάσεις δεδομένων. Αυτό ίσως περιπλέκει τα πράγματα, πάντως η εμπειρία μας έχει δείξει ότι μπορούμε να βοηθήσουμε και τη Δανία όπως και τις υπόλοιπες χώρες και τις διοκτικές αρχές. Με εξαίρεση την άμεση πρόσβαση στο σύστημα πληροφόρησης, γιατί αυτό είναι ένας νομικός περιορισμός που ισχύει και δεν μπορεί να έρθει. Εγώ νομίζω ότι απάντησα στις περισσότερε ερωτήσει. Να δώσω λίγο το λόγο και στον Φερνάντο όμως να απαντήσει πιο ειδικέ ερωτήσεις. Αν δεν απατώμα, έχουμε τέσσερα λεπτά. Επομένω, σύντομα θα προσπαθήσω να απαντήσω σε πιο συγκεκριμένε ερωτήσει. Ε, Μα ρωτήσατε για τις κυβερνοεπιθέσεις και ποιος είναι ο αριθμός τους. Διαπιστώνουμε ότι είναι μεγάλος, διαπιστώνουμε ότι είναι ένα φαινόμενο καθημερινό, επιχειρήσεις και άλλοι θεσμοί, θεσμικά όργανα ε, δέχονται τέτοιες επιθέσεις. Όσον αφορά την προστασία, δεν χρειάζονται μόνο τεχνικά μέσα, για την αντιμετώπιση των κυβερνοεπιθέσεων, αλλά επίσης είναι και ένα ζήτημα ε, εκπαίδευση, αν θέλετε. Βρίσκουν πάντα οι εγκληματίε τον πιο αδύναμο κρίκο. Επομένω, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια εκπαίδευση, μια κατάρτιση του προσωπικού. Συχνά διαπιστώνουμε ότι χρησιμοποιείται η κοινωνική μηχανική, χρησιμοποιείται η επαφή με συγκεκριμένα άτομα εντό μια επιχείρηση για να εισαχθεί malware, για παράδειγμα. Ε, η γνώση λοιπόν του προσωπικού για τα θέματα και η ευαισθητοποίηση του για τα θέματα τη κυβερνοασφάλεια είναι σε ορισμένε περιπτώσει ο πιο αδύναμο κρίκο. Χρειαζόμαστε λοιπόν και, τα, και την ευαισθητοποίηση και τα εργαλεία και επίση τα εργαλεία μετά για τη διερεύνηση. Ετέθη επίση ένα ερώτημα σε σχέση με την εκμετάλλευση παιδιών, τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών έχουμε μια καλή συνεργασία με όλα τα κράτη-μέλη. Και η καταπολέμηση της παιδικής εκμετάλλευσης είναι προτεραιότητα και στο, στη στρατηγική impact. Είναι δύσκολο βέβαια να έχει κανείς στατιστικά στοιχεία, ε, να γνωρίζει ακριβώς ποιες ήταν οι τα αποτελέσματα των διαφόρων ερευνών στις οποίες η Europol ε, υπάρχει υποστήριξη. Όμως, αν το δούμε συνολικά τα τελευταία 20 χρόνια, έχει υπάρξει μια αύξηση των, ε, των, ε, των ερευνών για τέτοιου τύπου περιπτώσεις. Ε, το deepfake, ναι, είναι μια νέα τεχνολογία η οποία αξιοποιείται από τους εγκληματίες. Για να σας δώσω κάποια πρόσφατα στοιχεία. Εμείς στη Europol συλλέγουμε στοιχεία από τις διάφορα εθνικά κέντρα για τα ε, ε, πιθανώς απαχθέντα παιδιά, για τα παιδιά που έχουν εξαφανιστεί. Και ε, προσπαθούμε να αποστείλουμε σε όλες τις χώρες ε, που συνεργάζονται, είναι 18, τα σχετικά στοιχεία. Φέτος είχαμε 300.000 τέτοιες αναφορές, το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να μιλάμε για πάνω από 300.000 θύματα. Προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε λοιπόν τα κράτη-μέλη να φιλτράρουν αυτές τις αναφορές. Δεν είναι όλες εξίσου σοβαρές στο ίδιο επίπεδο ποιότητας σε σχέση με τα στοιχεία που γνωρίζουμε. Και είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι στον τομέα αυτό χρειαζόμαστε περισσότερους πόρους, χρειάζεται να επενδυθούν περισσότεροι πόροι. γιατί χρειάζεται συνεργασία πολλών για να καταπολεμήσουμε το έγκλημα το σεξουαλικό που στρέφεται εναντίον των παιδιών και από την κοινωνία των πολιτών, όχι μόνο από τις διοκτικές αρχές για παράδειγμα και χρήσιμο θα ήταν σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υπάρχει ένας συντονισμός για την καταπολέμηση της παιδικής εκμετάλλευσης σε όλα τα επίπεδα. Ε, κάτι, κάτι τέτοιο φανταζόμαστε όταν μιλούμε για ένα κόμβο, για ένα hub, όχι αναγκαστικά υπό, υπό την Europol, αλλά είναι, είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια οργάνωση ομπρέλα που να συντονίζει τις πρωτοβουλίες στο, επίπεδο, στο τομέα αυτό. Στον τομέα λοιπόν της εκμετάλλευσης ανηλίκων, τι χρειάζεται, χρειαζόμαστε εργαλεία και χρειαζόμαστε και κατάρτιση για να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο. Ε, έχουμε στο πλαίσιο της Europol μια ομάδα εργασίας για την ταυτοποίηση θυμάτων. Συναντιόμαστε και επί δύο εβδομάδες αναλύουμε υλικό, ε, ε, βίντεο, φωτογραφίες, παιδικής εκμετάλλευσης και προσπαθούμε από κοινού να βρούμε ποια στοιχεία ποια μπορούν να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε ότι το έγκλημα διαπράχθη στην Ισπανία, στη Γαλλία, στη Γερμανία και μετά να ε, παράσχουμε τις σχετικές πρωτοβουλίες στις εθνικές ε, διοκτικές αρχές. Το σύστημα αυτό δεν μας βοηθάει μόνο να ταυτοποιούμε τα θύματα, αλλά επίσης είναι και ένας τρόπος ανταλλαγής εμπεριών. Ε, και κατάρτισης των αρμοδίων αρχών. Με αυτή την πρωτοβουλία όμως διαπιστώνουμε ότι καταφέρνουμε να αναλύσουμε μόνο ένα μικρό μέρος του υλικού που έχουμε στη βάση δεδομένων μας. Και όταν σας μιλώ για υλικό, ε, πρόκειται για εκατομμύρια αρχεία, τα οποία ακόμα δεν είχαμε τη δυνατότητα να αναλύσουμε εξαιτία αυτής της έλευσης πόρων. Όπως το είπε και ο συνάδελφος, λοιπόν, χρειάζεται ε, περισσότερη, χρειάζονται περισσότερες επενδύσεις στον τομέα αυτό, περισσότερη ανθρώπινη πόρη, περισσότερη κατάρτιση και περισσότερα εργαλεία. Αναφέρθηκε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι και η ανάπτυξη του συστήματος των ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στη Europol να λαμβάνει απευθείας αποδεικτικό υλικό από ιδιωτικού φορεί. Μέχρι στιγμή χρειάζεται πάντα να περάσουμε από τι εθνικέ διοκτικέ αρχέ και αυτό είναι ένα εμπόδιο. Ε, θα βοηθήσει να έχει περισσότερε δυνατότητε η Europol να λαμβάνει αυτό το αποδεικτικό υλικό κατευθείαν και μετά να το δημοιράζει στι υπόλοιπε αστυνομικέ αρχέ. Αυτά από την πλευρά μου. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε και τους δυο και τον αναπληρωτή επιχειρησιακό διευθυντή της Europol, τον κύριο Φαν Χέμερτ και τον συναδελφό του, Φερνάντο Ρουίθ. Σας ευχαριστώ επίσης που τους συναδέλφους που ρώτησαν, ε, έθεσαν τα ερωτήματά τους με τρόπο που θα μας επιτρέψει ακριβώς να κλείσουμε το θέμα αυτό στις 12.30. Βεβαίως θα συνεχίσουμε την συζήτηση μαζί σας και την δηλαδή απόψεων μου ζήτησαν οι συνάδελφοι αν θα μπορούσε να διανεμηθεί η έντυπη μορφή της έκθεσης για τις απειλέ σε όλα τα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Το... Η έκθεση Αιόκτα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να την εκτυπώσετε. Τώρα την παρουσίασή μου θα τη στείλω στη γραμματεία της Επιτροπής σας για να διανεμηθεί σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Προχωράμε. Συνεχίζουμε με το σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης. Το σημείο 10 αφορά τη θέσπιση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης. Αρμόδια εισηγήτρια είναι η κυρία Μίρια Μντάλη. Καλώς ήρθατε κυρία Ντάλη. Θα μας ενημερώσετε για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ε, για το κανονισμό που θεσπίζει το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης. Είχαμε δύο τριμερείς διαλόγους και στα λίγα λεπτά που έχω θα σας κάνω μια ενημέρωση για την κατάσταση. Στον πρώτο τριμερή διάλογο παρουσιάσαμε τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό, όπως επιβεβαιώθηκε και από την Επιτροπή μας και από την Ολομέλεια. Και μάλιστα η αλληλεγγύη, εξωτερική διάσταση, η δική στόχη του Ταμείου και η χρηματοδότησή του ήταν βασικές προτεραιότητες το θέμα της άμεσης ε, χρηματοδότησης τοπικές και περιφερειακές αρχές, πόροι για τη μετεγκατάσταση και την ε, επανεγκατάσταση, ε, επικοινωνία και κατεξοδότηση πράξη, βασικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο δεύτερο τριμέρι διάλογο σημειώσαμε κάποια πρόοδο σε διάφορα θέματα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το θέμα της αλληλεγγύης, του στόχου ταμείου, την αρχή της εταιρική σχέσης και την κατεπίγουσα αρρωγή. Πάντω το θέμα της αλληλεγγύης επισημάναμε ως πιο σημαντικό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για το θέμα αυτό έχουμε ευρία συνένεση σε, σε ολόκληρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο θεωρεί ότι είναι σημαντική αρχή η ε, αλληλεγγύη, αλλά θα πρέπει να συμπεριληφθεί ως βασικός στόχος, γιατί αν δεν αναφέρεται ως ειδικό στόχος η αλληλεγγύη του Ταμείου, θα έχουμε παλινδρόμηση σχέση με την παρούσα κατάσταση και θα συνεχίσουμε και στου επόμενου τριμερεί διαλόγου να επαναφέρουμε το θέμα τη αρχή αλληλεγγύη. Σε ό,τι αφορά του στόχου, έχουμε πέντε στόχου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το Ταμείο. Ένα από αυτού είναι η αλληλεγγύη και διαχωρίζουμε το θέμα τη νόμιμη μετανάστευση με την κοινωνική ένταξη. Το Συμβούλιο θέλει ω ειδικό στόχο την αλληλεγγύη και θέλουν το θέμα τη ε, νόμιμη μετανάστευση να συνδυαστεί με την ε, ένταξη. Επίσης, θα πρέπει να δούμε τι κονδύλια προβλέπονται για την νόμιμη μετανάστευση και για την ένταξη ξεχωριστά. Επίση, θα πρέπει να συνδέσουμε τους στόχους με το περιεχόμενο. αλλιώς δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε κατά, κατά πόσο το Ταμείο θέλει τους στόχου του σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση. Θέλουμε να αποφύγουμε ε, επικάλυψη με το άρθρο 6 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων. Η έκβαση ε, των, διαπραγματεύσεων για, το κοινό, για τον οργανισμό περί κοινών διατάξεων θα πρέπει να διαφυλάσει τις, ε, τους στόχους του Ταμείου Σύλλου και Μετανάστευσης. Επίσης, συζητήθηκε και η χρηματοδότηση των επιμέρους στόχων. Εμείς επιμένουμε ότι θα πρέπει να συμβάλλουμε με το Ταμείο στην υλοποίηση όλων μας των στόχων και προς και έχουμε ελάχιστα ποσοστά ε, δαπανών για τους στόχους. Το Συμβούλιο χάρη ε, ευελιξίας δεν θέλει τέτοια ελάχιστα ποσοστά, γιατί κατά τη γνώμη μας όμως τα ελάχιστα ποσοστά είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να αποδώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην υλοποίηση των στόχων του Ταμείου τα κράτη-μέλη. Επίσης, το θέμα της κατεπίγουσας ε, βοήθειας, της ε, έκτακτης αρρωγής. Πιστεύω ότι θα σημειώσουμε πρόοδο, αλλά θα πρέπει να συζητήσουμε και τη δυνατότητα παροχής της έκτακτης ενίσχυσης ε, από τους κεντρικούς φορείς που το έχουν ζητήσει. Και θα πρέπει αντίστοιχα να προβλέψουμε και προϋπολογισμό. Εγώ η συγγήτρια περιορίζομαι από την διαπραγματευτική εντολή που είναι βάση των διαπραγματεύσεων για μας και Στη διάρκεια των τριμερών διαλόγων ε, υπερασπίσαμε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που είναι πια γνωστή, δημόσια και πρόθεσή μου είναι να σημειώσω το δυνατό μεγαλύτερη πρόοδο στη διάρκεια της Φιλανδικής Προεδρίας, παρόλο που έχω επίγνωση ότι δεν είναι ξεχωριστό αυτό το θέμα του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευση από την υπόλοιπη συζήτηση για το ΠΔΕΛΤΑΠΗ. Σε μερικά σημεία έχουμε κολλήσει ή προχωρούμε σημειωτών ε, για θέματα που το Συμβούλιο δεν έχει εντολή. Έχουμε και τεχνικούς ε, τριμερείς διαλόγους. Η επόμενη, ο επόμενος τριμερής διάλογος θα γίνει ε, στο εγγύς μέλλον. Σας ευχαριστούμε κυρία Ντάλη που μας συνόψισατε τη μέχρι τώρα πρόοδο των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο. Θα ακούσουμε και τους κοιόδους ηγητές, αν επιθυμούν φυσικά να λάβουν το λόγο. Ο κύριος Λέναρς από το ΕΛΚ πρώτα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε κάτι οι ηγητές. Είμαστε στις διαπραγματεύσεις. Έχουμε κάποιες διαφορές σε θέματα περιεχομένου. Πάντως, ε, νομίζω πολύ σωστά έκανε την ε, σύνοψη των τριμερών διαλόγων η συγγήτρια. Ε, προσβλέπουμε συνέχιση των συζητήσεων και ελπίζουμε να έχουμε αίσιο, αίσια έκβαση στο μέλλον. Ο κύριος Χουκ από το Ρινίο, ο κύριος Μάρκερτ από τους Πράσινους. Θέλει κανείς να μιλήσει, δεν είναι υποχρεωτικό. Άμα θέλετε. Άμα επιμένετε να μιλήσω. Να συμφωνήσω με αυτό το οποίο είπατε. Χαίρομαι για το ότι συνεργαστήκαμε στενά στις διαπραγματεύσεις αυτές που δεν θα είναι εύκολες. Πρέπει να τονίσουμε ότι ο βασικός στόχος εδώ πέρα δεν είναι να χρηματοδοτούμε τρίτες χώρες, αλλά να στηρίξουμε ε, τα κράτη-μέλη για να επιδείξουν αλληλεγγύη στους ε, πρόσφυγες που έρχονται. Ευχαριστώ. Κύριο Σκόφοντ. Όχι. Κέμπα. Κύριε Χουκ. Εδώ είστε. Θέλετε να σχολιάσετε. Χωρίς μικρόφωνο. Να με συγχωρείτε που καθυστέρησα φαίνεται ότι ήρθε την κατάλληλη στιγμή, ως συνήθως. Ε, να πω κάτι, είναι πολύ σημαντική αυτή η νομοθεσία, να ευχαριστήσουν κυρία Νταλή, η οποία στις διαπραγματεύσεις εκπροσώπησε ολόκληρο το Κοινοβούλιο πάρα πολύ καλά. Και νομίζω μετέφερε τις θέσεις μας στο Συμβούλιο Κομισιόν, ε, ότι πόσο σημαντικό είναι δηλαδή να Έχουμε στήριξη ειδικά στην ένταξη και θέλω να τονίσω αυτήν την λέξη. Γιατί για την ομάδα μας το κομμάτι της ένταξης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι άνθρωποι έρχονται στην Ευρώπη ως πρόσφυγες πρέπει να ενταχθούν. Να μην είναι ξένοι που θα ζουν ανάμεσά μας, αλλά να έρθουν στις κοινότητές μας. Γιατί μιλάμε για παιδιά που θα πάνε στο σχολείο, οι ενήλικοι, θα μάθουν τη γλώσσα, ε, θα βρουν κάπου να δουλέψουν να είμαστε μια κοινωνία. Και επ' αυτού η ομάδα μας θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό η αλληλεγγύη του άρθρου 8 να τονιστεί. Η ομάδα μας λοιπόν αναμένει την επικοδομητική συνεργασία στον τρίτο γύρο διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Δεν βλέπω την κυρία Κέμπα. Δεν βλέπω τον κύριο Ορμπάν για την ΚΟΕ. Αν δεν έχει κάποιο άλλο να πει κάτι, μπορούμε να επιστρέψουμε νομίζω στην εισηγήτριά μας. Έχετε να πείτε κάτι? Όχι? Ωραία. Έχουμε ψηφοφορία την 11η πρωινή. Αλλά πρώτα απ' όλα να σας πω το χρονοδιάγραμμα. Όχι, όχι, όχι χρονοδιάγραμμα δεν έχει. περιμένουμε τις διαπραγματεύσεις, δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Υπάρχει και κάτι άλλο πριν το χρονοδιάγραμμα, το 11 έχει αναβληθεί. Έχει πάει για τις 5.30 το απόγευμα. Αυτό το οποίο αφορά την κυρία Φαγιών. Ο Ταμείο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης ε, Συνόρων. Δηλαδή, Έχουμε ψηφοφορία ηλεκτρονική. Στις 11. Στις 11. Διάλειμμα λίγων λεπτών. Λοιπόν, προτείνω γιατί αν το κάνουμε τώρα θα παραπονιούνται οι συνάδελφοι ότι δεν ε, το κάναμε την ώρα που ήταν προγραμματισμένο. Συμφωνείτε? Ναι. 11. Ναι, όχι. Όχι. 11. Διάλειμμα. Για να ψηφίσουμε 11 ακριβώς. Το πρωί, ε. 11 το πρωί. Μην φύγετε. Για να μπορέσουν να έρθουν και οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Αναλυτόρα. colleagues, Συνάδελφοι, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ που ήρθατε. Λοιπόν, σας περιμέναμε για να έρθετε 11 ακριβώς για την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Θα είναι σύντομη η ψηφοφορία μάλιστα και θα ολοκληρωθεί έτσι η σημερινή συνεδρίαση μέχρι τις 2.30 ε, που θα επαναλάβουμε. Με συνεδρίαση με τις επιτροπές ΝΤΕΒΕ ε, και γυναικών, αν δεν κάνω λάθος, στις 2.30 ώρα. Λοιπόν, σύντομη ψηφοφορία. Σχέδιο σύστασης της κυρίας Βυσνιεύσκα την οποία ευχαριστούμε. Το θέμα εδώ είναι να ψηφίσουμε την σύναψη πρωτοκόλλου με την Ελβετία και το Λιχτενστάιν. Για την εξέταση ετοιμάτων ασύλου στα κράτη-μέλη στην Ελβετία, για την πρόσβαση στην Eurodac, για σκοπούς επιβολής νόμου. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε. Μία τροπολογία. Μόνο. Και μετά ψηφίζουμε το σχέδιο σύστασης. Πρώτη ψηφοφορία αφορά την τροπολογία. Φροντίστε να είναι έτοιμες οι ηλεκτρονικές κάρτες, είστε όλοι στην θέση σας. Θα σας περιμένουμε κυρία Μελό. Έτοιμοι όλοι. Ψηφίζουμε την τροπολογία. Πάμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζουμε τη σύσταση, του κείμενο, του σχεδίου σύστασης ε, για τη συμφωνία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ε, μεγάλη πλειοψηφία. Θα τη δίναμε συγχαρητήρια αν ήταν εδώ. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.